Καλημέρα σας. Θα συνεχίσουμε τη συναισθήση της Επιτροπής μας με το σημείο 16 της ημερησίας διάταξης, πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής εξάπλωσης χωροκαταθεκτικών και εξωτικών ειδών. Όπως ξέρετε, τον ε, Σεπτέμβριο δόθηκε αυτή η γνωμοδότηση στον κύριο Ντέιβις, ορίστηκε ο κύριος Ντέιβις ως εισηγητής λοιπόν και σήμερα ακριβώς θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Ντέιβιτ. Παρακαλώ, του κύριου Ντέιβις, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν. Έχω υποβάλει ορισμένε τροπολογίε για την γνωμοδότηση και θα φροντίσω να είναι σχετικέ για αυτήν εδώ την Επιτροπή, μια και η Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι η αρμόδια. Σε γενικέ γραμμέ έχω καλύψει τι ε, γενικέ αρχέ που καλύπτουν ε, θέματα περιβαλλοντικά και του θελάσσιου περιβάλλοντο. Ε, Καταρχά όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ΓΔ περιβάλλοντος ε, και ιδιαίτερα σε, γενικά, σε γενικότερες γραμμές από την Επιτροπή. Μιλάμε για κάποια χωροκατακτητικά είδη και τις προτεραιότητες δράσης. Λέγεται ότι υπάρχουν 28 διαφορετικά χωροκατακτητικά ξένα είδη. αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και ο τρόπος που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα περιορίσει είναι τελείως ε, τεχνητός. Ε, κάποιο είδος ε, τα είδη που μπαίνουν στη λίστα αξιολογούνται σύμφωνα με το ε, πόσο σπάνια είναι, το οποίο θεωρούμε εμείς λάθος. Επίσης θεωρούμε λάθος το ότι όσο χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι μόνο εκείνα που βρίσκονται εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα μεταναστευτικά είδη που ε, μεταναστεύουν από βορρά προς νότο ενδεχομένως ε, να ε, είναι σε θέση να προκαλέσουν περιβαλλοντικές ζημιές και δεν είναι απαραίτητο να μεταναστεύουν δια της οδού, αλλά και δια της θαλάσσιας οδού. Αυτό που ζητώ εγώ είναι επαναθεώρηση των ε, περιορισμών και αξιολόγηση των ειδών βασισμένα στον κίνδυνο που ενδεχομένως να προκαλέσουν. Μετά από συστάσεις της ε, Γενικής ε, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος έχω ποσοτικοποιήσει την, τις προβλέψεις. Ε, θεωρούμε ότι η ποσοτικοποίηση των προβλέψεων πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να γίνονται με βάση το είδος και να υπάρχει μια ε, κατάλληλη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και των οικονομικών ε, συνεπειών. Και Αυτά τα χωροκατακτητικά είδη δεν είναι και σπάνια. Τα βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, στο, κανάλι που περνάει από την αυλή μου. Διάφορα είδη πανίδας και χλωρίδας. Και κανείς δεν ξέρει ποιες, είναι θα είναι οι περιβαλλοντικές συνέπειες και οι συνέπειες στα ενδυμικά είδη αυτών των χωρακατακτητικών ειδών. Έχω ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις στη διατύπωση σχετικά με τις αξιολογήσεις και όσον αφορά τους ε, τεχνητούς ε, περιορισμούς. Τέλος, ε, σε περίπτωση ειδών που είναι παρόμοια, δηλαδή το ίδιο είδος πουλιού, για παράδειγμα, με διαφορετικό χρώμα αυτερών. Αυτά τα είδη θα πρέπει να τα βλέπουμε ως ένα, ως μια οικογένεια ειδών και όχι ως ξεχωριστά είδη. Ιδιαίτερα εφόσον τα ίδια αυτά μπορούν να προκαλέσουν τις ε, ίδιες ε, ζημιές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντέιβις, η κυρία Πατράου, εκπροσωπώντας του κυρίου Κουν, γιατί ο κύριος Κουν απουσιάζει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως, παίρνω το λόγο εκ μέρους του κυρίου Κουν. Θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη για την απουσία του. Αλλά έχει μια πολύ σημαντική συνεδρίαση στην εκλογική του περιφέρεια σήμερα το πρωί, επομένω ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πρόταση αυτή. Και αναγνωρίζοντας ότι η αρμόδια επιτροπή είναι επιτροπή περιβάλλοντος, ε, η οποία δεν έχει ακόμη παρουσιάσει γνωμοδότηση, λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Κομισιόν Και βεβαίω απευθύνεται στον κύριο Ντέιβις που είναι ο εισηγητή αυτής της γνωμοδότηση για τη δική μας επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά του κύριου Ντέβις, λέει ότι συμφωνεί με τον κύριο Ντέβις για την τροπολογία του για το άρθρο 4, σημείο 4, να μην περιοριστεί ο κατάλογος των ειδών. Η ερώτηση στην Κομισιόν είναι ποιο είναι η αιτιολόγηση για το νότο των 50 ειδών. Ο κύριος, ο κύριος Κούν υποστηρίζει την τροπολογία του εισηγητή για την υποβολή εκθέσεων στο άρθρο 19.1β για τη συμπερίληψη των θαλασσίων υδάτων η δημιουργία μια ομάδα επιστημονικών συμβουλών, τροπολογία για το 21α, επίσης υποστηρίζεται από το σκιώδη του ΕΛΚ. Οι ανησυχίες ε, του σκιώδους εισηγητή είναι το άρθρο 23, δηλαδή η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν. Στο άρθρο 4 η Κομισιόν θα έχει την αρμοδιότητα να υιοθετήσει και να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των χαρακτηριστικών ξένων ειδών μέσω εκτελεστικών πράξεων και στο άρθρο 23 την αρμοδιότητα να υιοθετήσει εξουσιοδότηση πράξης. Αυτή η ανάθεση αρμοδιοτήτων ε, διευκρινίζεται σε ένα συγκεκριμένο άρθρο και η επιστημονική συμβουλή σχετίζεται με το άρθρο όπου περιγράφονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να μπουν αυτά τα είδη στον κατάλογο. Ο σκιωδής εισηγητής του ΕΛΚ πιστεύει ότι η ανάθεση εξουσιών στην Κομισιόν μέσω των εκτελεστικών πράξεων καθώς και η ανάθεση μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της πρότασης. Θα ήθελε μια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία για το θέμα αυτό της ανάθεσης αρμοδιοδίτων στην Κομισιόν για αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία ή για τα μη ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης, αν πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που έχουν ουσιαστική ή μη ουσιαστική φύση. Και αυτή είναι η συνεισφορά του αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πατράου. Εξ ονόματος του κυρίου Κούν, η κυρία εξ του κυριου κουν η κυρια λοβιν Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα. Εμείς οι πράσινοι συμφωνούμε απόλυτα με την προσέγγιση ότι τα, ο κατάλογος των 50 ειδών είναι τελείως ανεπαρκής. Θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε δει τις ε, τεράστιες ε, συνέπειες ε, με τα νερά τα οποία χύνουν τα πλοία και μέσω αυτών ε, ξένα είδη έχουν ε, βρεθεί στην Βαλτική και όχι μονάχα εκεί αλλά σε όλα τα είδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το τραγικό παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας ε, όπου ένα είδος μέδουσας έχει, jellyfish, έχει εξαφανίσει διάφορα είδη και ήδη γίνεται και κάτι τέτοιο στην Βαλτική θάλασσα. Επίσης, έχουμε τις κλιματικές αλλαγές που θα επηρεάσουν ε, την διάδοση ειδών, ξένων ειδών. Θα υπάρξει μια διαταραχή, αν θέλετε, στην γεωγραφική εξάπλωση των ειδών. Ε, επομένως ε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τον συγκεκριμένο κατάλογο ειδών. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν παγωμένο κατάλογο. Πρέπει ε, να αναθεωρείται, να εξετάζουμε κάθε είδος ξεχωριστά και υποστηρίζουμε την διαγραφή του περιορισμού στα 50 είδη. Επίσης υποστηρίζουμε την ιδέα ότι δεν είναι μόνο τα εξοκοινωτικά είδη τα οποία μας απασχολούν Προφανώς, εάν ε, μεταφέρουμε και στο ιστορικό της ευρωπαϊκής κοινότητας κάποια ίδια από ένα σημείο στο άλλο που δεν ανήκουν, προφανώς θα υπάρχουν ε, ε, συνέπειες και, και στα ενδυμικά είδη. Επίσης, όσον αφορά την τις ποσοτικές προβλέψεις, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσουν τα ξένα είδη. Μπορεί να γίνει κάποια, κάποια στιγμή και σε κάποιο επίπεδο, αλλά από οικονομικής πλευράς δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου προβλέψεις ποσοτικές από τα king crabs, από τα, μεγάλα καβούρια τέλος πάντων, δεν ξέρω τι οικονομικές συνέπειες μπορεί να αντλήσουμε. Μπορεί να καταστρέψουν και το οικοσύστημα ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και θα υποβάλουμε και κάποιες ε, τροπολογίες έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε την προσπάθειά του. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, παρακαλώ. Thank you, Chair. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση σήμερα. Διαβάσαμε την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Ντέιβις με μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα περιέχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα εστιάσουμε σε ορισμένες από αυτές, ε, διότι τις θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές. Ο κύριος ε, Ντέιβις και ορισμένοι από τους συναδέλφους του ανέφεραν το όριο των 50 ειδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτήθηκε ποιο είναι το σκεπτικό και η λογική πίσω από την επιλογή των 50 ηθών ε, εν ώψη των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και η εξήγηση είναι η εξή. Καταρχά, το όριο των 50 ειδών ήταν ε, προορισμένο να εφαρμοστεί σε, πρώτη, σε πρώτο στάδιο. Σχεδιάστηκε για να δώσει την ασφάλεια στο αρχικό στάδιο, στα κράτη-μέλη, του ότι ο αριθμός αυτός δεν θα ξεπεραστεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν περισσότερο ακριβείς υπολογισμούς. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα που ήθελα να τονίσω. Δεύτερο θέμα και επίσης πολύ σημαντικό είναι το εάν κάποιο είδος είναι ενδυμικό σε ένα μέρος ε, της Ευρώπης αλλά χωροκατακτητικό σε κάποιο άλλο σημείο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την απειλή ε, των ειδών και δεν το κάνουμε. Αντίθετα πιστεύουμε πως είναι πάρα πολύ ε, σημαντική η απειλή. Όμως το να εστιάσουμε σε ήδη ε, ξένα προς την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι που αποφασίσαμε λόγω της ανάγκης ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα και το σύστημα που έχουμε εφαρμόσει έχει σχέση και συνδέεται με την, ευρωπαϊκή, με την εσωτερική αγορά σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τώρα, όσον αφορά το αν κάποια είδη είναι ενδημικά σε ένα μέρος της Ευρώπης αλλά προκαλούν ζημιά σε κάποιο άλλο, είναι σημαντικό και το αναγνωρίζουμε αυτό. Και να σας πω όλες ότι το θέμα αυτό συζητείται σε πεδομάδων ομάδων εργασίας στο Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σκοπεύουμε να ασχοληθούμε ένεργα με το θέμα αυτό. Έχουμε τώρα κάποιες ανησυχίες σχετικά με το σύστημα των ε, εξαιρέσεων και των παρεκκλήσεων, διότι ανησυχούμε για ενδεχόμενη μείωση της προστιθέμενης αξίας και προσπαθούμε να εξετάσουμε το θέμα δίνοντας έμφαση στο περιφερειακό στοιχείο και δίνοντας ε, έμφαση σε ορισμένα κράτη-μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα από αυτά τα χωροκτητικά είδη. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση και καλωσορίζουμε την ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Άγγνου και ξέχασα να του το δώσω. Παρακαλώ. Μην ανησυχείτε, Πρόεδρε. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο ζούμε σε ένα νησί και αυτό μας δίνει κάποιες ευκαιρίες, κάποιες δυνατότητες. Ο τρόπος ε, που το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό είναι ότι όλες αυτές τις διαφορετικές χώρες τις θεωρήσαμε μία και αυτό αναγκάζει το Ηνωμένο Βασίλειο. να δείτε το θαλάσσιο, το ναυτιλιακό παράδειγμα, ε, τα ε, τα πλοία μας ε, ουσιαστικά είναι αργά και έχουμε και εμείς προβλήματα με τα χωροκατακτητικά ίδια, αλλά τα προβλήματα μας μπορεί να μην είναι τα ίδια, ε, γιατί εμείς... Ο σκίουρος είναι ε, στην κορφή του καταλόγου μας και θα θέλαμε να αναλάβουμε μέτρα γι' αυτό, αλλά δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να υποστηρίξω να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό στη χώρα μου. Νομίζω ότι εμείς θα έπρεπε να το κάνουμε, να επιλέξουμε εμείς το είδος που θέλουμε να θέσουμε σε προτεραιότητα και να επιλέξουμε και την ταχύτητα με την οποία θέλουμε να κινηθούμε. Ευχαριστώ κύριος Ντέβις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Άγνους για τη συνεισφορά του γιατί φέρνει και στην Επιτροπή εδώ τις συζητήσεις που έχουμε συνεχώς στο Ενωμένο και νομίζω ότι τονίζει την πραγματικότητα της ε, κατάστασης ε, που είναι ε, πάρα πολύ απομακρυσμένη. Ναι, πράγματι η χώρα μου είναι νησί και αυτό δίνει ένα πλονέκτημα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτών των χωροκατακτητικών ειδών. Είναι χιλιάδες τα αυτά. Είναι αδύνατο να σταματήσουμε την εξαπλωσή τους και το ότι είμαστε νησί δεν έχει διαφορά γιατί είμαστε τμήμα της Ευρώπης και του κόσμου. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό και ε, φυσικά δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που να μας εμποδίζει να πάρουμε μέτρα ε, σε σχέση με το σκύρο και να προστατεύσουμε τους εναπομείνατες ε, κόκκινους ε, σκύρους και να ε, μπορέσουμε να σταματήσουμε την εξάπλωση του Αμερικανικού σκύρου αλλά χρειαζόμαστε και διεθνή συνεργασία, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία στην περίπτωση αυτή, γιατί έχουμε συλλογικέ εμπορικέ συμβάσει και μέσω του εμπορίου και των εμπορικών διευθετήσεων εξαπλώνονται πολλά από αυτά τα είδη. Και άκουσα και τη λέει Κομισιόν. Φυσικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν μπορούμε να πάμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να πάμε πάρα πολύ μακριά και αν ε, φυσικά θέλουμε αποτελεσματικά μέτρα θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν ε, τα κατάλληλα μέτρα για να προσπαθήσουν να σταματήσουν την εξάπλωση των ειδών αυτών που θα έχουν προσδοριστεί ως είδη που ήταν σοβαρό κίνδυνο όμως ε, απλώς ε, δεν μπορεί να βάλει κανείς ε, αυτούς τους περιορισμούς. Εμείς θα θέλαμε φυσικά να πούμε στα κράτη-μέλη «Α, μόνο 50 ήδη μας ανησυχούν», αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανείς, γιατί δεν στέκει επιστημονικά. Και Φυσικά η Κομισιόν πολύ σωστά στην έκθεσή της μας είπε ότι χρειάζεται πρώιμη δράση και η πρόληψη μπορεί να είναι πολύ καλή από άποψη εξοικονόμησης χρημάτων. Αν καθυστερούμε, σημαίνει, και θα επανέλθω στους κύρους, και να σας υπενθυμίσω ότι δεν λάβαμε δράση κατά του Αμερικανικού σκύρου και έτσι τώρα οι αυτόχθονες σκύρου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε κίνδυνο. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν για τα επιχειρήματα αυτά αλλά ε, θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι σκόπιμο αυτό το τεχνητό όριο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντέιβις. Να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών ε, είναι στις 4 Δεκεμβρίου, το 12 το μεσημέρι. Και αν δεν υπάρχει Κάποιο άλλο σχόλιο, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 17, Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλικού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευση, έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση φυλάκων για το προσωπικό των ελευτικών σκαφών. Πρόκειται για μια σύμβαση του 1995. Η σοσιαλιστική ομάδα είχε αναλάβει την γνωμοδότηση αυτή και η κυρία Τομάκ είναι εισηγήτρια και αρμόδια επιτροπή είναι επιτροπή απασχόληση Τώρα, όπως και την στο προηγούμενο σημείο θα ακούσουμε την παρουσίαση της πρότασης εκ μέρους ε, της Κομισιόν καταρχήν και θα προβούμε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μετά την κυρία Τομά. Να ακούσουμε την Κομισιόν. Ο κύριος Γκαλιτσιόλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη παρουσίαση της πρότασης αυτής. Τα κράτη-μέλη θα επικυρώσουν ή θα υπογράψουν τη, Διεθνή τη Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ε, ε, για τα πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών που έχουν ε, υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον Άιμο να σας ενημερώσω για το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής και τον λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη πρέπει να πρέπει, ενθαρρύνονται μάλλον να επικυρώσουν ή να υπογράψουν αν δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Η σύμβαση αυτή οθετήθηκε το 1995 αλλά τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου του 2012. Ένα χρόνο μετά την ε, επικυρίωση από το 15ο κράτος. Εμείς είμαστε, είμαστε παρατηρητές στην ΆΙΜΟ. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι της σύμβασης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 1978, αν επιτρέπετε, όταν η ΆΙΜΟ υιοθέτησε μία σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης και έκδοσης πιστοποιητικών ε, για τους ναυτικούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια, αν θέλετε, των ε, θαλασσίων ε, επικοινωνιών. Το 1994 υιοθετήθηκε μια οδηγία του Συμβουλίου η οποία έχει ενημερωθεί και έχει τροποποιηθεί, έχει γίνει και ένα recast εντωμεταξύ και από την 35, από την οδηγία 35-2012 τροποποιήθηκε για άλλη μια φορά. Το 1978 δεν υπήρχε ε, ακόμα δεν υπήρχαν οι ορισμοί τους οποίους ε, χρειαζόμαστε, γιατί τότε δεν, δεν αντιμετώπιζα με το θέμα ε, με τέτοιους σφαιρικούς χαρακτήρες. Και ε, ο κανονισμός που αφορούσε τους ε, ναυτικούς δεν συμπεριλάμβανε τους αλείς. Αργότερα υιοθετήθηκε ένα νομικό κείμενο για τους αλείς και είναι μια απλουστευμένη μορφή της σύμβασης που αφορούσε τους ναυτικούς. Αφορούσε τα αλληλευτικά σκάφη πάνω από 25 μέτρα και κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Τους skippers, ε, ε, τους αξιωματικούς, τον καπετάνιο δηλαδή, τους αξιωματικούς, τους ε, υπαξιωματικούς και τον ασυρματιστή. δεν υπήρχαν δεν, υπήρχαν, δεν είχαν συμπεριληφθεί συγκεκριμένα επαγγέλματα. Η σύμβαση αυτή όριζε ελάχιστα, ελάχιστες προδιαγραφές, κατάρτιση και η ιατρική φροντίδα. Βέβαια, καλό είναι τα, τα πρότυπα αυτά και οι προδιαγραφές αυτές να ολοκληρωθούν, να βελτιωθούν. Το 1995 πάνω από 20, από 20 κράτη υπέγραψαν τη σύμβαση, τέσσερα μόνο την επικύρωσαν και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε, στην διαδικασία ε, ολοκλήρωσης της επικύρωσης. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω ότι άλλα κράτη όπως το Μαρόκο, η Μαυριτανία, το Κυριμπάτι έχουν ήδη επικυρώσει τη σύμβαση αυτή και αναφέρω εδώ τώρα τρία κράτη με τα οποία έχουμε διμερείς αλληλευτικές συμφωνίες. Η Κομισιό επέστησε την προσοχή στους, ε, στους ε, υπουργούς ε, αλληλείας ότι χρειάζεται επιγόντως να επικυρωθεί η σύμβαση αυτή είναι θέματα... Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι αρμόδιοι υπουργοί, γιατί είναι και θέματα εκπαίδευσης, παραδείγματο χάρη. Ε, υπάρχουν, κράτη όπου ο αρμόδιος για τα θέματα λίας δεν είναι και αρμόδιος για θέματα της εκπαίδευσης. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υπογράψουν αν δεν ή να επικυριά επικυρώσουν αυτά που δεν έχουν επικυρώσει. 22 σας είπα έχουν υπογράψει για κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες Είπαμε ότι ε, ε, μιλάμε για συγκεκριμένα επαγγέλματα και για συγκεκριμένα μεγέθη. Άρα είναι ένα μικρό κομμάτι ε, του αλλιευτικού στόλου, του κοινοτικού αλλιευτικού στόλου. Τα πιστοποιητικά αναφέρονται σε συγκεκριμένα προσόντα και μόνο από τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, μόνο κάποια ε, εκδίδονται με βάση το IMO και επιτρέπουν ε, να εργάζονται ε, οι ναυτικοί πάνω στα συγκεκριμένα αλληλευτικά σκάφη. Καλό θα είναι δηλαδή να πρέπει φροντίσουμε έτσι ώστε το, όλο το πλήρωμα να κατέχει αυτού του είδους τα πιστοποιητικά. Τώρα, στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων έχουμε την οδηγία 2035-36 που αναθεωρείται και η νέα εκδοχή θα δημοσιευθεί σύντομα γιατί υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η οδηγία αυτή προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την κατάρτιση και την εμπειρία και ε, επιτρέπει να ε, γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στα διάφορα επαγγελματικά προσόντα και στα επαγγέλματα. Άρα ένας εργαζόμενος από ένα κράτος μέλος, ο οποίος θέλει να εργαστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, το φιλοξενών ας πούμε κράτος μέλος, όπου εκεί το επάγγελμα αριθμίζεται από εθνική νομοθεσία ή από την πρακτική, θα πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε τα προσόντα και αν τα προσόντα είναι ίδια, τότε επιτρέπεται να εργαστεί αυτός ο εργαζόμενος ε, στα αλληλευτικά σκάφη του φιλοξενούντος, ε, της φιλοξενούσας χώρας. Άρα σύμφωνα με τον κανονισμό, με τη σύμβαση, δεν χρειάζεται συγκεκριμένο πιστοποιητικό, διότι η φιλοξενούσα χώρα ε, είναι υποχρεωμένη να συγκρίνει τα προσόντα και αν δεν είναι αντίστοιχα τα προσόντα, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος να ε, κάνει μια συμπληρωματική κατάρτιση ή εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσει να εργαστεί. Επομένως η έλλειψη πιστοποιητικού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού δεν απαγορεύει στον εργαζόμενο να δουλέψει σε ένα ξένο αλληλευτικό σκάφος διότι ε, ε, ε, ε είμαστε μέσα σε μια ενιαία αγορά. Επομένως, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, τους δοθεί η άδεια να επικυρώσουν, διότι μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην ε, σύμβαση με του ΙΣΑΙΜΟ και τον ε, μηχανισμό τον ευρωπαϊκό, ο οποίος δεν απαιτεί συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Επομένως, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση και ταυτόχρονα να υποβάλουν μια ε, επιφύλαξη ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, προέχει η, ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με την σύμβαση, διότι δηλαδή δεν μπορούν να επιβάλλουν ε, ένα επιστοποιητικό άιμο ε, σε μια χώρα που ακόμα δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όπως σας είχα πει, τέσσερα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει μέχρι στιγμής. Επομένως, ε, για το σχέδιο ε, προβλέπει ότι τα κράτη αυτά θα πρέπει να ε, εκφράσουν μια επιφύλαξη. Δηλαδή υπογράψαμε, επικυρώσαμε στη σύμβαση, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στις σχέσεις των κρατών μελών, για τα επαγγελματικά προσόντα η ευρωπαϊκή νομοθεσία προέχει. Ε, κανένα άλλο σχόλιο. Στο άρθρο 3 προβλέπουμε την επικύρωση μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό τώρα πλέον δεν είναι ρεαλιστικό, διότι η στέρηση επομένως προβλέπουμε μια άλλη διαδικασία που θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θεωρηθεί η απόφαση. Τέλος πάντων, ε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Τώρα θα δώσω το λόγο στην συγκίτρια, κυρία Τωμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, όντω η θέση σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι η σύμβαση αυτή υπεγράφει το 1995 και τέθηκε σε ισχύ το 2012, εξηγείται επειδή χρειάζονταν 15 κράτη να έχουν κυρώσει και ο ρυθμός αυτός πληρώθηκε το 2012. Τα κράτη-μέλη δεν ε, επιτρεπόταν ε, να επικυρώσουν ε, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια σύμβαση που έχει πολύ αξιόλογους στόχους γιατί θέλει να βελτιώσει την κατάρτιση των αλλιέων και να το πω και αυτό ότι η ε, αλληλείς είναι οι τελευταίοι στους ε, οποίους ε, δίνουμε προτεραιότητα σε σχέση με θέματα κατάρτισης, γιατί είναι πιο παλιές οι συμβάσεις. Έτσι λοιπόν είναι πολύ καλός ο σκοπός, η βελτίωση της κατάρτισης κυρίως για την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια των ναυτικών και την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και την ασφάλεια ε, σε σχέση με τα ατυχήματα για να αποφευθεί η ρήπανση στη θάλασσα. Επίσης, ένας άλλος σημαντικός στόχος ε, είναι η εναρμόνιση των προσόντων. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Και επίσης, ε, και να πω και εγώ, όπως και εκπρόσωπος της Κομισιόν, ότι όλα αυτά δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα. Ωστόσο, θα έχουμε βέβαια και την δυνατότητα να το συζητήσουμε, απλώς εκφράζω κάποιες σκέψεις εδώ. Παραμένει λοιπόν, όπως έλεγα, ότι το, το κύριο πρόβλημα το οποίο ε, είναι ε, τα σκάφη άνω των 25 μέτρων. Ε, ξέρουμε ότι ε, είναι ένα πολύ μικρό μέρος ε, του Ευρωπαϊκού Στόλου και τα σκάφη ε, κάτω των 45 μέτρων για τις περιορισμένες ζώνες. Αυτό μας εκπλήσει κάπως, όμως, όπως και να έχει, έχουμε τα μικρά σκάφη ε, τα οποία δεν εξυπηρετούνται όπως πρέπει ως προς τις απαιτήσει και αν δούμε τις στατιστικά στοιχεία θα δούμε ότι αυτά που πλήττονται περισσότερο δεν είναι τα σκάφη των 45 μέτρων ενώ ε, στην ε, ε, αλία βλέπουμε ότι είναι διαδεδομένα τα ατυχήματα και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και κυρίως τα σκάφη κάτω των 25 μέτρων. Επομένως θα πρέπει να προβληματιστούμε για το ζήτημα αυτό. Αναφέρεται ότι υπάρχει, υπάρχουν σκάφη πάνω των 25 μέτρων, περιορίζονται 45 μέτρα περιορισμένα και μετά έχουμε τα μεγάλα σκάφη. Και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα σκάφη δεν έχουμε κανέναν ορισμό. Είναι κάποια ερωτηματικά λοιπόν που ίσως θα έπρεπε να τεθούν. Και να σας πω ότι επειδή δεν γνωρίζω πολύ καλά τη διαδικασία, τι θα κάνουμε, θα γνωμοδοτήσουμε ή υπέρ κατά. Δηλαδή, θα είμαστε υπέρ ή κατά και δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή εκτός αν ανεπίσημα έλθετε να συζητήσουμε πριν τη σύνταξη της έκθεσης για να μπορέσετε να μου υποβάλλετε τις παρατηρήσεις που θεωρείτε σκόπιμες. Και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνταξη της νομοδότησης στις 7 Δεκεμβρίου, με παρουσίαση στην Επιτροπή 22-23 Ιανουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή αλληλιά το Φεβρουάριο και στην Ολομέλεια το αργότερο το Μάρτιο. Άννα... Ε, φυσικά μπορέσει και η Κομισιόν να διατηρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα, γιατί και αυτή πρέπει να εκπονήσει γνωμοδότηση. Μάλιστα, κύριε Πατρά. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για αυτό το έγγραφο. Θα ήθελα λοιπόν να πάρω το λόγο. Εγώ νομίζω ότι για τη σύμβαση αυτή η σύμβαση αυτή είναι κάτι πολύ σημαντικό και σε σχέση με το θέμα της αναγκαιότητας να επιτραπεί στα κρατημέλη να υπογράψουν, τα είπε η Όμως η αλεία στη θάλασσα είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Και πολλές φορές συμβαίνουν ατυχήματα ε, που μπορεί να είναι και θανατηφόρα και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουμε, έχουμε ε, σε όλο τον κόσμο 24.000 ε, θανάτους αλλιέων. Δηλαδή πρόκειται για ένα κλάδο με πολύ ψηλό κίνδυνο. Επομένως, ε, στον κλάδο της ελίας έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο το 7% των θανατηφόρων ατοχημάτων και 2,4% περισσότερες φορές είναι υψηλότερος ο κίνδυνος στον κλάδο της αλίας για να συμβούν ατυχήματα. Αυτό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς ε, εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Στον τομέα της αλίας, εγώ θα έλεγα ότι πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα οικονομικής επαγγελματικής δραστηριότητας, ο κίνδυνος του ατυχήματος φαίνεται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, σαν να είναι ουσιαστικά κάτι εγγενές ε, του επαγγέλματος ε, και αυτό είναι λυπηρό και θα πρέπει να συζητηθεί και να καταπολεμηθεί σε οργανωτικό επίπεδο οι κύριοι παράγοντες κλειδιά που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τα εργατικά ατυχήματα σχετίζονται πάρα πολύ με την απουσία κατάρτισης ε, σε θέματα ασφάλειας ε, στο χώρο εργασίας και υπερβολική ανοχή στον κίνδυνο και ακριβώς ε, και για αυτούς ε, τους λόγους ε, έχουμε και μεγαλύτερο κίνδυνο στον τομέα της αλίας. Εγώ νομίζω ότι η κατάλληλη κατάρτιση είναι θεμελιώδης για να μειώσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων και διαπιστώνω ότι αναγνωρίζεται από την πολιτική στον τομέα της αλίας ότι χρειάζεται πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας και σίγουρα αυτές τις στοιχείες θα πρέπει να τις θέσουμε σε εφαρμογή από το 2014 μέχρι το 2020. Στο πλαίσιο αυτό το ίδιο το Ταμείο Αλίας αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα για να βελτιώσουν ε, τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας επί του σκάφους και να συμπεριληφθεί και η κατάρτιση ε, των ναυτικών και των αλλιέων και σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να αλλάξει η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα στον αλλιευτικό τομέα. Αν ε, ε, αναγνωρίσουμε τα προσόντα και προσδώσουμε επαγγελματική κατάρτιση, τότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μειωθούν τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα. Θα δούμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια της θάλασσας, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ε, και επομένω πρέπει αυτέ οι διατάξει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Εγώ νομίζω ότι όλοι εμείς δεν διαφωνούμε εδώ και η Κομισιόν αλλά και η Συγήτρια όπως και εγώ από την πλευρά του ΕΛΚ όλοι εμείς συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητη η σύμβαση και πήγουσα. Και εδώ αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι οι πτυχές που αναφέρει η κυρία Τομά αλλά να δούμε και ποιε πτυχέ θα μπορούσαν ε, να βελτιωθούν. Αν και βέβαια έχουμε θέμα αρμοδιότητα εδώ για να το πράξουμε αυτό. Πάντω, όπω και να έχει, αξίζει τον κόπο να υπογραμμίσουμε τουλάχιστον αυτές τις ανησυχίες ε, γιατί θέλουμε να γίνει ένα βήμα προς τα μπρο με ε, την έγκριση αυτή που ήδη έχει καθυστερήσει. Έτσι, λοιπόν, θα έπρεπε τουλάχιστον η σύμβαση αυτή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κλάδου όσο το δυνατόν περισσότερο. Επομένως, εγώ εδώ συμφωνώ με όσα υπόθηκαν από την εισηγήτρια την κυρία Τωμά. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τωμά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να ε, επικυρωθεί αυτή η σύμβαση, αλλά να επωφεληθούμε κιόλα για να υπογραμμίσουμε την ύπαρξη κάποιων προβλημάτων ε, κάποιων προβλημάτων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούσαμε για ε, πλοία λιγότερα των 24 μέτρων και συνέχεια υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα σκάφη, διότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα σκάφη αυτά. Δεν υπάρχει συνομιλητής για να συζητήσουμε το ε, σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν τα σκάφη κάτω των 24 μέτρων γι' αυτό καλό θα είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε, να διευκρινίσουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σκάφη τα μικρότερα των 24 μέτρων να επιμείνω ότι είναι τα σκάφη στα οποία έχουμε τα περισσότερα επαγγελματικά ατυχήματα, εκεί η μεγαλύτερη θνησιμότητα, είναι τα περισσότερα, τα περισσότερο ευάλωτα. και δεν είναι και ένοχα, αν θέλετε, για, όσον αφορά την θαλάσσια μόλυνση, αν μη τι άλλο. Υπάρχουν προβλήματα, βέβαια, αλλά για τους αλληλείς και για τους ναυτικούς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων και δεν τους καλύπτει η σύμβαση αυτή και ίσως θα μπορούσαμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, διευρύνουμε τη σύμβαση αυτή, να συμπεριληφθούν ε, και τα σκάφη τα μικρότερα των 24 σκαφών. Βέβαια πάντα για τα κοινοτικά αλληλευτικά σκάφη μιλάμε. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι. Όπως είπε και η κυρία Τόμα, 20 με 22 Ιανουαρίου θα γίνει παρουσίαση τη νομοδότηση, 17-18 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και θα πάει και στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Παρουσίαση από το θεματικό τμήμα των ενημερωτικών σημειωμάτων, αποδοτικότητα του ελευτικού στόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επιδοτήσει για τα κάρσιμα στο ελευτικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση από του Γερμάρτισον και Αλεσάνδρα Μπορέλ, προσώπων του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Εγώ νομίζω ότι χωρίς χρονοτριβή να τους δώσουμε το λόγο για να μας παρουσιάσουν ε, αυτά τα ενημερωτικά σημειώματα. Και θα συνεχίσει ο κύριος ε, Αντιπρόεδρος με την Προεδρία. Okay, good morning. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δύο αυτές μελέτες που ζητήσατε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για, τις, για τα θαλάσσια θέματα. Το όνομά μου είναι Γιάν Μάρτινσον και ε, συνεργάστηκα με την Αλεσάνδρα Μπορέλο και πριν από την Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τις εσωτερικές πολιτικές. Πριν προχωρήσουμε στην ουσία της έκθεσης, να πούμε δύο λόγια για τον εαυτό μας, για να ξέρετε ποιοι είμαστε. Ε, είμαστε από τη Γενική Διεύθυνση που, ε, στην οποία ανήκει το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Ασχολούμεθα με την αλία κυρίως, αλλά και με τα ναυτικά θέματα, φιλιακά θέματα εν γέννη. Το κέντρο ερευνών είναι, αν θέλετε, το εσωτερικό επιστημονικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ε, δίνουμε συμβουλές ε, επικεφαλής προφανώς είναι ο κύριος Μπαρόζο, η επίτροπος ε, είναι η κυρία Μαϊρέ Γκόγκενχαμ Κουίν, γενικός διευθυντής ο Ντομινίκ Κριστόρια, αλλά ο οποίος θα πάει τώρα στην έρευνα. Όπως σας είπα, το βασικό μας ε, θέμα, η βασική μας καθήκον είναι να προσφέρουμε επιστημονική συμβουλή, σε επιστημονικές συμβουλές σε, όλες, σε όλα τα σε όλους τους τομείς ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Εμείς ε, ε, προσφέρουμε συμβουλές στον τομέα της αλληλείας. Συνεργαζόμαστε και με άλλες γενικές διευθύνσεις. Δεν ασχολούμεθα μόνο με την αλληλεία αλλά και την αυτιλιακή κίνηση, τα ατυχήματα, επίβλεψη και επιτήρηση ναυτιλιακή. Ο στόχος μας και οι στόχοι μας και τα καθήκοντά μας είναι ευρύτερα. Έχουμε μία προσέγγιση πολύπλευρη, τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφόρησης, συλλογή ε, ε, δεδομένων, προωθημένες ε, και προχωρημένες τεχνολογίες, ε, γενετική και γενόματα, τα οποία θέλαμε να ε, συμπεριλάβουμε και στην διαχείριση της αλληλείας και και το 2012 είχαμε παρουσιάσει κάποια εργασία μας, ίσως να το θυμόσαστε, ίσως και όχι. Όπως σας είπα, θέλουμε, ο βασικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε επιστημονική υποστήριξη στον τομέα της αλληλείας συνεισφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερο στην μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και βοηθάμε έτσι ώστε να έχουμε μια βιώσιμη αλληλεία, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και ε, προβλήματα όπως ας πούμε η διατροφική ασφάλεια η διαφάνεια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, κυρίως σε σχέση με αυτά τα οποία θα σας πει η κυρία Μπορέλο σε λίγο. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, συμμετέχει ιδιαίτερα και πολύ, πολύ κοντά στην εργασία της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συλλέγει τα δεδομένα τα οποία προσφέρουν τα κράτη-μέλη, τα ε, προωθούμε στην Επιστημονική Επιτροπή Αλίας και ενημερώνουμε τους επιστήμονες και προσφέρουμε επιστήμονες στην Επιτροπή αυτή. Βλέπετε, έχουμε την ε, ετήσια έκθεση για την αλληλεία είναι ένα από τα, μία από τις δημοσιεύσεις μας. Επίσης, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ε, την διάδοση των δεδομένων και των πληροφοριών σε όλους τους ε, ενδιαφερόμενους, ας πούμε στην Επιτροπή Αλίας, αν ενδιαφέρεται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας και το λέω αυτό διότι εάν δείτε την ε, συλλογή των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, project μας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Αυτή η μελέτη την οποία ζητήσατε δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί πριν από μερικές δεκαετίες. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, π.χ. ας πούμε η έλλειψη δεδομένων. Άρα, αλλά όμως να τονίσω ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για, την, ε, για το μέλλον της αλίας. Όπως σας είπα επίσης, κάνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την αλληλεία. Σας ανέφερα και την ετήσια έκθεση, αλλά και ε, την ε, προσοχή μας σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο και Θέλουμε να δούμε και πώς, είναι οι, πώς λειτουργούν οι επιτροπές στις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η ιδιατοκαλλιέργεια θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Λοιπόν, η Αλεσάνδρα Μπορέλο τώρα θα σας παρουσιάσει τις μελέτες που είχετε ζητήσει για την αποδοτικότητα του ελευτικού στόλου και για τις επιδοτήσεις για τα κάθισμα στον ελευτικό τομέα. Όταν μας, δώσατε τις, μας αναθέσατε τις εκθέσεις αυτές, πρέπει να σας πω ότι θεωρήσαμε ότι ήταν τεράστιο το έργο, γιατί δεν θα είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Υπάρχουν κάποια κενά βέβαια. Ε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε όμως, έτσι αυτό θεωρήσαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Ποπέσκου που μας υποστήριξε τα θέματα επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατόπιν ε, τούτου θα δώσω το λόγο στην αδελφό μου την Αλεσάνδρα Μπορέλο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών. Ας αρχίσουμε με την ε, αποδοτικότητα και του εμπορικού λευτικού στόλου. Είναι μια συνολική αξιολόγηση με ανάλυση που έγινε σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο τομεακό. Έπειτα, παρέχουμε πληροφορίες για την κερδοφορία του αλευτικού ε, στόλου στο σημείο αναφορά 2. Έπειτα, μας ζητήθηκε να παρέχουμε μια γενικότερη αξιολόγηση της ε, συνεισφοράς του αλληλευτικού τομέα την ε, εγχώρια καθαριστή παραγωγή. Αυτό έγινε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, κάναμε μια ανάλυση της, ε, των οικονομικών ενισχύσεων στον ευρωπαϊκό αλληλευτικό τομέα. Η ανάλυση μας βασίστηκε στα δεδομένα που μας παρήχαν τα κράτη-μέλη, τα οποία συλλέχθηκαν μετά από, την, ε, από την ε, ζήτηση του 2013. Εμείς συμπληρώσαμε τις πληροφορίες ε, που μας έστειλαν τα κράτη-μέλη κατόπιν του αιτήματος του 2013 με ε, δεδομένα από ενδιάμεσες αξιολογήσεις και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Ελίας. Η ανάλυση μας εστίασε στα δεδομένα που μας έστειλαν τα κράτη-μέλη. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που είχαμε ήταν από το 2011. Εδώ βλέπετε την κάλυψη των δεδομένων. Όπως βλέπετε, δεν είχαμε δεδομένα για την Ελλάδα και είχαμε μερική κάλυψη όσον αφορά την Ισπανία και την Κύπρο. την Εστονία. Εδώ βλέπετε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο. Το 2011 ο Ευρωπαϊκός Αλλιευτικός Στόλος αριθμούσε 65.000 σκάφη. Δεδομένου όμως ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ε, δεν ε, συνυπολογίστηκαν, Ο αριθμό αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 76% του συνόλου των αλληλευτικών ε, σκαφών. Χωρητικότητα σε τόνου ήταν 1,64 εκατομμύρια και 5,9 εκατομμύρια κιλοβάτ του στόλου. Τα σκάφη αυτά είχαν συνολικά 3,8 εκατομμύρια ημέρες στη θάλασσα. Όμως να επαναλάβω ότι τα δεδομένα αυτά είναι ελλειπή. Εδώ βλέπετε Ποιού δείκτε χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε την ε, αποδοτικότητα και την απόδοση του στόλου. Χρησιμοποιήσαμε ε, ακαθάριστο περιθώριο κέρδους, καθαρό περιθώριο κέρδους και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του στόλου, το εισόδημα μάλλον του στόλου, ε, ενέρχεται σε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με κόστος 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η καθάριστη προστιθέμενη αξία ανήλθε στα 3,4 δισεκατομμύρια και όπως βλέπετε μόνο 5 κρατημέλη, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία ε, κάλυψαν 80% του της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Εδώ είναι τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης κερδοφορία του αλληλευτικού στόλου σε επίπεδο κρατών μελών. Γενικότερα ο Ευρωπαϊκός Αλληλευτικός Εκλάδος το 2011 έχει ακαθάριστη προσθέμενη αξία στο 48% του ε, συνολικού ΑΕΠ και περιθώριο ακαθάριστου κέρδους 18%. Περιθώριο καθαρού κέρδους ήταν 6% και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε πόσο ο Ευρωπαϊκός Αλληλευτικός Στόλος ήταν κερδοφόρος στο διάστημα αυτό. Αυτό βασικά είναι βασισμένο στα στατιστικά στοιχεία που είχαμε και που ήταν αξιόπιστα, το οποίο δεν κάλυπταν όλα τα κράτη-μέλη. Παρατηρήσαμε σε τέσσερις χώρες ε, αρνητικό καθαρό περιθώριο κέρδους σε, για 8 χώρες τα ποσοστά ήταν σχετικά ουδέτερα και σε 5 χώρες τα ποσοστά ήταν, κέρδους ήταν υψηλά. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης που έγινε σε επίπεδο τομέων. Εδώ ε, βλέπουμε ότι το 2011 ε, η, τα σταθερά αλληλευτικά εργαλεία ήταν περισσότερο κερδοφόρα από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι από ό,τι τα υπόλοιπα και από ό,τι πελαγότρατες. Αυτό βέβαια πρέπει να το αναλύσουμε Έχοντα υπόψη ότι ορισμένα αλληλευτικά εργαλεία ήταν περισσότερο κερδοφόρα σε κάποια κρατημέλη από ό,τι σε κάποια άλλα. Είναι λοιπόν μια πολύ γενικότερη αξιολόγηση αυτή και συνολική. Το TOR 3 τώρα είναι μια ανάλυση της ε, συνεισφοράς του αλλιευτικού κλάδου στο ΑΕΠ. είδαμε ότι το 0,03% είναι το ποσοστό συνεισφοράς του ευρωπαϊκού στόλου σε εθνικό επίπεδο. Σχεδόν για όλα τα κράτη-μέλη η εκαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν στο 2,5% του συνολικού ΑΕΠ με μία εξαίρεση. διεξήχθη μια παρόμοια ανάλυση όπου συγκρίναμε ε, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον αλληλευτικό και στον αγροτικό τομέα. Εδώ είδαμε ότι ο αγροτικός τομέας ήταν περισσότερο κερδοφόρος με μερικές εξαιρέσεις. Να σας πω όμως ότι ο... ότι τα στατιστικά αυτά στοιχεία και τα νούμερα αυτά είναι πιο γενικά. Εάν εξετάσουμε επιμέρους κάποιες ε, παράκτιες ε, περιοχές θα δούμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Μια πρόσφατη ανάλυση που έγινε για αυτές τις περιοχές ε, έδειξε ότι σε 25 μέρη της Ευρώπης η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της αλίας είναι πάνω από 10% του, της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται στις περιοχές αυτές και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έπειτα, μας ζητήθηκε να παράσχουμε πληροφορίες όσον αφορά την συνεισφορά, την οικονομική συνεισφορά στην ε, συνολικότερη αλληλευτική πολιτική. Η κύρια συνεισφορά λοιπόν στον ε, αλληλευτικό κλάδο προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας ε, στο χρονικό διάστημα 2007-2013. Υπήρχαν και άλλες ε, οικονομικές ενισχύσεις, τις οποίες ε, δεν αναλύσαμε στην μελέτη μας. Όπως για παράδειγμα διάφορες φορολογικές ελευθερίνσεις ε, για τα καύσιμα και και η de minimis aid. Χρησιμοποίησαμε δεδομένα όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις του αληφτικού στόλου από το 2011. Έπειτα συμπληρώσαμε τα στατιστικά μας στοιχεία με βάση τον άξονα προτεραιότητας 1 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Λίας 2007-2013. Αυτές οι δύο πηγές που χρησιμοποιήσαμε είναι συμπληρωματικές στην μελέτη μας, έχουν όμως αναλυθεί με διαφορετικό τρόπο, διότι υπάρχουν επικαλύψεις. Και ο, η μία μέθοδος επιτρέπει αναλύσεις σε, εθνικό επίπεδο και επίπεδο κλάδων, ενώ η όχι. Επίσης, είδαμε ότι οι άμεσες ενισχύσεις εισοδήματος ήταν πάνω από 98 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και αυτές οι ενισχύσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τράτες και από σκάφη που χρησιμοποιούσαν ε, παθητικά λεφτικά εργαλεία και ήταν μέχρι 12 μέτρων. Αυτό ήταν στο περί... στο 5% του συνολικού εισοδήματος. Βέβαια υπάρχει διαφορά απλώς όσον αφορά την χρήση των ε, επιχορηγήσεων αυτών. Αυτό που είδαμε επίσης ήταν ότι η κερδοφορία με ή χωρίς επιχορηγήσεις και συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που είχαμε δεν είχε μεγαλές διακυμάνσεις για του, τον ε, αλλιευτικό κλάδο. Εδώ βλέπετε ορισμένα παραδείγματα αυτού, αλλά μπορείτε να βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες στην ίδια τη μελέτη. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πηγή πληροφοριών, είδαμε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τον πρώτο άξονα του Ταμείο Αλίας ήταν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που αντιστοιχεί στο 1 τρίτο του συνολικού κονδύλου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας 2007-2013 και ήταν το υψηλότερο σε εθνικό επίπεδο. Είχε προγραμματιστεί για την Ισπανία, ακολουθώντας η Πολωνία και η Ιταλία. Ωστόσο, για όλες σχεδόν τις χώρες, το μερίδιο μεταξύ του μέσου προϋπολογισμού του προγράμματος και της ακαθάριστης ε, αξίας ε, για τον κλάδο, προσθέμενης αξία για τον κλάδο, ήταν κατώτερο από το 50%. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις είδαμε ότι ήταν υψηλότερο. Εδώ συνοψίζω τα όσα είπα για τους, ε, τη συγγραφή υποχρεώσεων υπαριθμών 1. Εδώ ο στόλος περιλαμβάνει 65.000 σκάφη, απασχολεί 127.000 αλείς και το 2011 παρήγαγε 3,5 εκατομμύρια εκφορτώσεις και 4,9 δισεκατομμύρια εκφορτώσεις. Ε, το περιθώριο κέρδους ήταν αρνητικό μόνο για τα σέρα κράτη-μέλη, καθάριση προσωπική εξής σε εθνικό επίπεδο είναι συνήθως κάτω του 0,2% του εθνικού ΕΠ, ενώ ε, έχουμε 0,03% συνήθως και οι άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις είναι κάτω του 5% για τους περισσότερους τόλους για το συνολικό εισόδημα και 1% για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο, ορισμένα, μόνο τμήματα του στόλου ε, θίγησαν σοβαρά σε σχέση με το ε, περιθώριο ακαθάριστου κέρδους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα θέλετε να απαντήσετε ερωτήσεις τώρα ή προτιμάτε να προχωρήσετε στην επόμενη έκθεση. Υπάρχουν κάποια μέλη της Επιτροπής τα οποία θα ήθελα να κάνουν ερωτήσεις για αυτό τώρα. Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη. Okay. So, this is the terms of reference for εδώ έχουμε τη συγγραφή υποχρεώσεων για τη δεύτερη μελέτη. Εδώ θα δούμε τα φορολογικά επιδόματα για τον ε, ευρωπαϊκό τομέα κλάδο αλίευσης. Κατόπιν θα αναλύσουμε το επίπεδο των φόρων για τον κλάδο αν ε, δεν υπήρχαν ε, αυτά τα επιδόματα για τα καύσιμα. Κατόπιν ε, θα δούμε ποιο είναι το εισόδημα που έχουν χάσει οι κυβερνήσεις λόγω σε αυτές τις φοροαπαλλαγές και θα συγκρίνουμε τα διάφορα τμήματα του στόλου σε σχέση με το πόσο εξαρτώνται από την κατανάλωση καυσίμων για να αξιολογήσουμε το ωφέλη για τους διάφορους στόλους που προέρχονται από αυτά τα φορολογικά επιδόματα, της φορολογικής ελαφρύνσης και κατόπιν μας ζητείτε να δούμε, να κάνουμε μια εκτίμηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τον Ευρωπαϊκό Στόλο και να συγκρίνουμε αυτή την κατανάλωση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε πάρα πολλές πληροφοριών Κύριε, ήταν μια έκθεση ερευνητική που ε, ε, παρουσίασε ο Οργανισμός Συνεργασίας και Αναπτύξης ΟΣΑ. Επίσης, ε, πήραμε στοιχεία από τον ΟΣΑ και από, την Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και επίσης κάναμε και μία μελέτη και χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες ειδικών φόρων κατανάλωσης ε, που έχει δημοσιεύσει η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ταξούντ μαζί με τα κράτη-μέλη. Και για την άλλη έκθεση χρησιμοποιήσαμε στοιχεία που μας έστειλαν τα κράτη-μέλη τύπου TCF και δεδομένα από τη Eurostat. Εδώ για κάθε πηγή πληροφοριών βλέπετε ποια συγγραφή υποχρεώσεων ε, έχει χρησιμοποιηθεί. Παρουσίασα ήδη τη διαφάνεια αυτή, αλλά και εδώ η κάλυψη δεν ήταν ε, πλήρης. Λοιπόν, για τη συγγραφή υποχρεώσεων υπαριθμών 2, ε, εδώ βλέπετε το ιστορικό από το 2003 1993 δηλαδή τα κράτη-μέλη θα δεν θα επιβάλλουν φορολογία για ενεργειακά προϊόντα που ε, παρέχονται ως καύσιμα για στόχους πλοήγησης εντός κοινοτικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της αλίας. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της ανάλυσής μας προέκυψε ότι σχεδόν όλες οι χώρες, ε, ο τομέας δηλαδή ο κλάδος της αλίας εξαιρείται 100% από την καταβολή φόρων για τα καύσιμα με την εξαίρεση έξι κρατών μελών, Εστονία, Λιθουανία, Πορτοκαλία, Ελλάδα, κάτω χώρες. Για τη Βρετανία είναι μερική η απαλλαγή αυτή και κάναμε μία σύγκριση με λίγες χώρες ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ε, αναμένεται είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χώρες για τις οποίες δεν δίνονται επιδοτήσεις για τα καύσιμα στον τομέα της έλίας, ενώ σε άλλες χώρες συμβαίνει το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα τη συγγραφή που χρειάζεται παρθούν δύο. μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε ποιο θα ήταν το επίπεδο των φόρων για τους αλείς, αν δεν υπήρχαν αυτά τα επιδόματα. Και εδώ παρουσιάζουμε το εθνικό ποσοστό φόρων για τον ντίζελ. Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2003-96 τα κράτη-μέλη έπρεπε να θέσουν ε, μία τιμή για το φόρο που να είναι υψηλότερη από την ελάχιστη αξία που είναι 330 ευρώ για χίλια λίτρα. Έτσι λοιπόν ε, βλέπετε ότι ενώ κάποιες χώρες μένουν πάρα πολύ κοντά στο ελάχιστο, σε αυτήν την ελάχιστο ποσοστό. Κάποιες ε, άλλες χώρες έχουν ε, θέσει ένα φορολογικό συντελεστή που είναι σχεδόν ο ε, διπλάσιος από την ελάχιστη τιμή. Μας ζητήθηκε λοιπόν να εκτιμήσουμε τα διαφυγόντα εισοδήματα για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω αυτών των φορολογικών επιδομάτων, των φορολογικών ελαφρύσεων. Και είδαμε ότι χάθηκε 1,05 δισεκατομμύριο ευρώ αναχρόνο και αυτό αντιστοιχεί στο 0,022% του συνολικού ευρωπαϊκού εισοδήματος. Σε εθνικό επίπεδο συνήθως για όλες τις χώρες ήταν κάτω του 0,2% του εθνικού εισοδήματος. Στη συνέχεια, συγκρίναμε τα διάφορα τμήματα του στόλου ανάλογα με την εξάρτησή τους από την κατανάλωση καυσίμων και υπολογίσαμε τους διάφορους δείκτες και παρουσιάζουμε τώρα εδώ μόνο ένα από τους δείκτες που υπολογίσαμε την ε, κατανάλωση καυσίμων ανά ημέρα στη θάλασσα. Όπως ε, βλέπετε, τα κινητά αλλιευτικά εργαλεία εξαρτώνται περισσότερο από την κατανάλωση καυσίμων ε, φυσικά όπως αναμένεται σε σχέση με τα στατικά, με τα σταθερά εργαλεία και είχαμε παρόμοια αποτελέσματα και όταν ε, συγκρίναμε το κόστος ε, του καυσίμου με το συνολικό επιχειρησιακό κόστος και είδαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις είναι ψηλότερο ακόμη και κατά 40% αλλά είδαμε ότι για το ίδιο τμήμα του στόλου και πάλι μπορεί να συμβεί το εξή. Ο ίδιος δείκτης να έχει εντελώς ε, διαφορετική τιμή από μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να είναι διαφορετικά, να διαφέρουν. Και φυσικά μπορεί να διαφέρει και το μεγέθος ε, του τμήματος του στόλου που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αν και πρόκειται για το ίδιο τμήμα του στόλου. Έτσι λοιπόν αυτά πρέπει να αναλυθούν λεπτομερέστερα για να έχουμε πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Τέλος, συγκρίναμε την κατανάλωση των καυσίμων σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεται για όλες τις άλλες χρήσεις ε, και είπαμε ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,22%. Εδώ χρησιμοποιήσαμε στοιχεία του 2009 για να φτάσουμε σε αυτό το μέσο όρο, γιατί δεν έχουμε πάντα πλήρη δεδομένα για την ε, κατανάλωση καυσίμων. Σε εθνικό επίπεδο ήταν ε, πάντοτε κάτω του 1,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Όταν ε, κάναμε σύγκριση με τον τομέα της γεωργίας, είδαμε ότι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάναμε στο 9,94% το μερίδιο αυτό, ενώ σε εθνικό επίπεδο συνήθως ε, ήταν κάτω του 30%. Εδώ βλέπετε και μία σύνοψη της έρευνας. Είδαμε λοιπόν ότι σχεδόν ε, σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει συνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρων καυσίμων. Φυσικά εδώ μιλάμε για τον κλάδο της αλίας. Βέβαια αυτό δεν ισχύει 100% για 6 χώρες και οι φορολογικοί συντελεστές για τα καύσιμα γενικά διαφέρουν ανά κράτος αυτό που πρέπει λοιπόν ε, να πληρώσουν ε, οι αλείς ε, χωρίς αυτήν την απαλλαγή επικύλη και το διαφυγόν εισόδημα είναι το 0,022% του ευρωπαϊκού εισοδήματο. Συνήθως τα σκάφη που χρησιμοποιούν ενεργά εργαλεία εξαρτώνται περισσότερο από τα καύσιμα, καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα Επομένως μπορούν να ωφεληθούν τα μάλα από αυτή την φοροαπαλλαγή και ο ελευτικός τομέας συνήθως καταναλώνει κάτω από 1% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, πολύ, κύριε Μπορέλο, για την παρουσίασή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν. Δεν κατάλαβα καλά το γιατί περίπου έξι κράτη-μέλη, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν περίπου μερική απαλλαγή για τα καύσιμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης η οποία δεν έγινε μόνο από εμάς. Εμείς χρησιμοποιήσαμε ε, τα στοιχεία που υπάρχουν στην έκθεση του ΟΑΣΕ και εμείς κάναμε μια πολύ σύντομη μελέτη, όμως όταν την ε, υποβάλαμε λάβαμε απάντηση μόνο από μερικές χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Σουηδία. Δεν νομίζω πως λάβαμε καμία απάντηση από τους εμπειρογνώμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί ήταν και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα στο οποίο έπρεπε να απαντήσουν. Δεν ξέρω ακριβώ τι έχει γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις νομίζω οι κάτω χώρες είχαν εξαίρεση για ορισμένους ε, τύπους ε, καυσίμων, για ντίζελ για παράδειγμα από φορολογία. Το πετρέλαιο δεν εξαιρούταν. Επίσης τα εσωτερικά ύδατα και τα παράκτια ύδατα αποτελούν μέρος της εξαίρεσης και όχι για παράδειγμα σκάφη του, της ανοιχτής θάλασσας. Μπορώ να σας δώσω βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες των Ηνωμένων αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά νομίζω πως ε, ε αν ε, στο παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, η μία χώρα, έχει, ε, μία χώρα εξαιρείται και η άλλη όχι, υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Επίσης, αυτό που ονομάζουμε κόκκινο ντίζελ ε, απολαμβάνει φορολογικών ε, ελαφρύνσεων, εξαιρείτε. Και αν ε, σε πιάσουν να χρησιμοποιείς αυτό το κόκκινο ντίζελ, όχι στα αγροτικά σου μηχανήματα, όχι στο τρακτέρ, αλλά στο αυτοκίνητο, έχεις πρόβλημα. Αλλά ίσως έχετε δίκιο, όταν, αν κάποιος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί κυροζίνη ή κάποιο άλλο είδος ε, πετρελαίου, πρέπει να πληρώσει φόρους. Λοιπόν, μου ζητήσετε δεδομένα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Συνολικές εξαιρέσεις καυσίμων για χρήση σε σκάφη εκτός από σκάφη που πλέουν σε εσωτερικά ύδατα. Δηλαδή υπάρχουν εξαιρέσεις για όλα τα σκάφη εκτός από εκείνα που πλέουν σε εσωτερικά ύδατα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει μερική εξαίρεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και να έχει όλες οι λεπτομέρειες των ευρημάτων μας βρίσκονται στους πίνακες 9 4 για εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Για την Πορτογαλία συγκεκριμένα βρήκαμε ότι οι εξαιρέσεις υπήρχαν για πετρέλαιο που χρησιμοποιείται σε σκάφη που πλέουν παράκτια και σε εσωτερικά ύδατα, όχι δηλαδή για τα σκάφη ανοιχτή θάλασσα. Και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι, υπήρξαν και, ότι υπήρξε και ένας εμπειρογνώμονας για την Πορτογαλία συγκεκριμένα, ο οποίος ε, παρήχε κάποια στατιστικά στοιχεία και βοήθεια, κάποια πρόσθετη έρευνα. Δηλαδή, για τον, δηλαδή ο στόλος ανοιχτής θάλασσας της Ισπανίας εξαιρείται ενώ της Πορτογαλίας όχι. Αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Θα αρχίσετε πόλεμο μου φαίνεται. Αλλά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Η κυρία Λόβιν. Όχι, ο κύριος Άγνιου. Πραγματικά συναρπαστική ήταν η παρουσίαση και Πολύ ωραία μας την παρουσιάσατε και μας δώσατε πολλές χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες δεν θα ξεχάσω. Το κόκκινο ντίζελ που χρησιμοποιείται στη Γεωργία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι ξέρετε 100%. Νομίζω πως ξέρετε μερικώς. Υπάρχει ένα... Υπάρχει λοιπόν αυτή η μερική εξαίρεση γι' αυτό και δεν μπορούσατε να μας δώσετε το πράσινο χρώμα στην, στον πίνακα αλλά το κόκκινο. Κοιτάξτε, Νομίζω ότι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση και τα οποία ίσως να χρήζουν περαιτέρω μελέτης, διότι εμείς συλλέξαμε κάποια στοιχεία και από άλλες πηγές. Δεν είναι αντικείμενο δικής μας ανάλυσης όλο το περιεχόμενο. Τέλος πάντων, λέει ο Πρόεδρος, νομίζω ότι τίθενται κάποια ενδιαφέροντα ερωτήματα για τον ανταγωνισμό. Κύριε Λόβιν, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για τις μελέτες. Όντως, ε, καλό είναι που έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Δεν κατάλαβα όμως ε, πολύ καλά στην πρώτη παρουσίαση όταν μιλήσατε για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τις επιδοτήσεις. Συμπεριλάβατε το διαφυγόν κέρδος ε, τον ε, για, τα, για τις επιδοτήσεις, για, τα, για τις ελαφρύνσεις, για τα καύσιμα στο θέμα, στα θέματα της κερδοφορίας. Στην πρώτη μελέτη, όχι, όχι, εννοώ γενικά, γενικά, όλες οι αναλύσεις που κάναμε για την πρώτη μελέτη, κυρίως όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες, στηρίχθηκε σε, στα δεδομένα από την Τράπεζα Δεδομένων. Για το... Και αυτή η Τράπεζα Δεδομένων αναφέρεται σε στοιχεία που αφορούν τις άμεσες επιδοτήσεις, ε, τις εισοδηματικές επιδοτήσεις. Κάποιες χώρες συμπεριλαμβάνουν τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα και άλλες χώρες δεν συμπεριλαμβάνουν τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα. Επομένως, δεν μπορώ να σας ε, ε, δώσω μία απάντηση άμεση. Επίσης ανέφερα ότι πέρυσι τον Απρίλιο οργανώθηκε ένα εργαστήρι στο Σαλέρνο της PG Econ που είναι μια υποομάδα αν θέλετε που ασχολείται με οικονομικά θέματα και εκεί ε, κατάρτισαν, εκπώνησαν ένα πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος και που αναφέρονται λεπτομερείς πληροφορίες ανά χώρα. Για κάθε χώρα μπορείτε να δείτε τι συμπεριλαμβάνεται στις άμεσες ε, εισοδηματικές επιδοτήσεις και τι δεν συμπεριλαμβάνεται. Κυρία Λόβεν, άρα η συνεισφορά του αλληλευτικού στόλου, αν θέλετε, για, την, για το συνολικό ε, ΑΕΠ της κοινότητας είναι 0,03% ενώ ε, για τις για τις ε, ε, φορολογικές ελαφρύνσεις, οι, ε, λαμβάνοντας υπόψη φορολογικές ελαφρύνσεις, η συνεισφορά του ελευτικού στόλου στην ενέργεια όλης της κοινότητας είναι 0,2%. Ξέρετε γιατί έχουμε αυτές τις φορολογικές ελευθερίνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι στην Ισλανδία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκείνοι πληρώνουν ε, τα καύσιμα κανονικά και τη φορολογία για τα καύσιμα. Αν θυμάμαι καλά, κάποια, υπάρχει κάποια συμφωνία του IMO. Δεν θυμάμαι καλά, θα μπορούσα να μας το διευκρινίσετε. Τι κρύβεται πίσω από, αυτή την, ε, από αυτές τις ελαφρύνσεις. Α, και άλλη μια ερώτηση Στον πίνακα 4 της μελέτης αναχώρα για την εκτίμηση του διαφυγόντος ε, των ε, εισοδήματος ε, αναχώρα είδα ότι για κάποιες χώρες πήγε για την Ιταλία έχει ένα διαφυγόν εισόδημα 362 εκατομμύρια ευρώ κατέτος. Τρελά ποσά. Και αν το συγκρίνετε ας πούμε με την Ισπανία που έχει 71 εκατομμύρια σε σχέση με τα 362 στην Ιταλία και η Ισπανία είναι πιο μεγάλο αλληλευτικό κράτος. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εξήγηση. 241 εκατομμύρια η Γαλλία, ας πούμε. διαφυγών εισόδημα που οφείλεται στις αυτές τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Λοιπόν, εάν συγκρίνουμε τους διάφορους τόλους, τα ποσά αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Η Δανία ξέρουμε ότι είναι για τα πελαγικά η δύναμη μεγάλο κράτος και έχει μονάχα 47 ε, εκατομμύρια διαφυγών ε, ε, εισόδημα. Έχετε κάποιες εξηγήσεις για τα ποσά αυτά και αν κατακλείδη. Σαν σχόλιο, αλλά καλό είναι να το δούμε, για τα σταθερά εξαρτήματα, το σταθερό εξοπλισμό, που για τις περισσότερες χώρες είναι ο πλέον επικερδής, χωρίς επιδοτήσεις, εξαρτάται λιγότερο από, την, από τα καύσιμα. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε πώς εξηγούνται αυτά τα τεράστια ποσά για κάποιες χώρες. Λοιπόν, να μας πείτε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές ανάμεσα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις κάτω χώρες που έχουν τεράστια διαφυγόντα εισοδήματα λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό πώς εξηγείται. Εξηγείται από το ο, του στόλο, χρησιμοποιούν περισσότερο σταθερά ή κινητά ε, εξοπλισμό, τι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ε, του διαφυγόντου εισοδηματός βασίζεται βασικά σε δύο τεινά στην ε, κατανάλωση καυσίμων σε εθνικό επίπεδο και το συντελεστή της φορολογικής απαλλαγής που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση δεν χρησιμοποιήσαμε για όλες τις χώρες τον ίδιο συντελεστή. Εκεί μάλλον οφείλεται η διαφορά, δηλαδή επειδή οι κανονικοί άνθρωποι πληρώνουν μία τιμή για τα καύσιμα και οι μία άλλη τιμή. Όμως χρησιμοποιήσαμε μία εκτίμηση που βασιζόταν σε στοιχεία τη εκθέση του ΩΣΑ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχαμε και περαιτέρω στοιχεία από τους εμπειρογνώμονε. Και όταν δεν είχαμε στοιχεία να χρησιμοποιήσουμε, θεωρήσαμε ότι ο συντελεστής, ο φορολογικός ε, συντελεστής, είναι αυτός που χρησιμοποιείται κανονικά για τα καύσιμα. Επομένως, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών σε σχέση με το συντελεστή που χρησιμοποιείται, όμως το κύριο ζήτημα είναι η συνολική κατανάλωση καυσίμων. Για τις πρώτες χώρες που έχετε εδώ, είχαμε πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμων καθόλου το έτος. Αλλά πήραμε το μέσο όρο από την, για την περίοδο 2002-2011. Και να σας πω ότι για κάποιες χώρες είχαμε όλα τα στοιχεία για όλη την περίοδο 2002-2011, ενώ για άλλες χώρες είχαμε τα τελευταία μόνο χρόνια. Επομένως, Καθώς η κατανάλωση καυσίμων μειώνεται σε πολλά κρατημέλη, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως για κάποιες χώρες για τις οποίες είχαμε πιο πρόσφατα στοιχεία να υπήρχε υποεκτίμηση της κατανάλωσης, ενώ για άλλες χώρες όπως η Ιταλία αξιολογήθηκε η πραγματική κατανάλωση, τα πραγματικά στοιχεία που μας είχαν δώσει. Περισσότερο δηλαδή εξαρτάται από την κατανάλωση καυσίμων. Γιατί όπως είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια για το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε πολύ υψηλό συντελεστή, φορολογικό συντελεστή για τα καύσιμα, ενώ εδώ δεν έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα από τα πρώτα κράτη σε σχέση με το διαφυγόν εισόδημα. Επομένως, η κατανάλωση είναι το στοιχείο που μετράει περισσότερο. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την κυρία Λοβίν. Και για τους κανόνες ε, του IMO, Δηλαδή, γιατί έχουμε αυτή την οδηγία της ε, φοροαπαλλαγής για τα καύσιμα. Απάντηση, η οδηγία ουσιαστικά εισήχθη το 2003. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι ο στόχος ήταν να βοηθήσει τους αλείς να προσαρμοστούν στις ε, αλλαγές, ε, στις διακυμάνσεις, στις τιμές των καυσίμων. Γιατί στη Γεωργία που είναι ο άλλος τομέας ο οποίος ε, λαμβάνει πολλές επιδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τέτοια απαλλαγή. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη ποιος είναι ο κύριος λόγος. Παρακαλώ κύριε Φράγα. Εμένα με εντυπωσιάζει όταν λέτε ότι στην περίπτωση της Ισπανίας ε, ότι ε, έχουμε εξαίρεση για όλο το στόλο σε σχέση με την καταβολή φόρου για τα καύσιμα. Στην πρακτική όμως, στην πράξη όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί όταν ε, μιλάμε για το στόλο ανοιχτής θαλάσσης, μεγάλων αποστάσεων, η κατανάλωση αυτών ε, των καυσίμων ε, γίνεται εκτός της Ισπανίας. Επομένως μπορεί να υπάρχει ένα στόλο στον Ινδικό ωκεανό ή στον Ειρηνικό ωκεανό μπορεί να περάσει και δύο-τρία χρόνια χωρίς να επιστρέψει στην Ισπανία. Επομένως, ναι, νομικά μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Και η απόδειξη είναι ότι όταν ε, ήρθε, παραδείγματος χάρη, ο στόλος, έχουμε το θηνελευτικό στόλο, ο οποίος ακριβώς ε, παραπονιέται για αυτά τα θέματα σε σύγκριση με το τι συμβαίνει με τρίτες χώρες. Ε, γιατί ε, ακριβώς καταναλώνουν αυτά τα καύσιμα όχι, εκτός της Ισπανίας. Δηλαδή, υποτίθεται ότι στην Ισπανία όλος ο στόλος λαμβάνει επιδοτήσεις, όμως τελικά αυτό δεν ισχύει για το στόλο μακρινών αποστάσεων, γιατί καταναλώνει τα καύσιμα εκεί όπου αλλιεύει. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε εκεί υπόψη, γιατί στην πράξη αυτά δεν ισχύουν, παραδείγματο χάρη για αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του στόλου που σα ανέφερα. Απάντηση. Πολύ καλό είναι που γίνονται όλα αυτά τα σχόλια. Ουσιαστικά για το ίδιο πράγμα, για την ε, φορολογική απαλλαγή. Όπως σας είπα, είμαι σίγουρη ότι πρέπει να ερευνηθούν πάρα πολύ τα θέματα αυτά, γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλές εξαιρέσεις και πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς ως ερευνητές. Γιατί το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, κυρίως αν λάβουμε υπόψη και την πίεση του χρόνου, το καλύτερο που μπορέσαμε να κάνουμε ήταν να οργανέσουμε τις πληροφορίες που είχαμε δει στη διάθεσή μας. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα σας μάλλες λέτε και θα έπρεπε να ερευνήσουμε εις βάθος το θέμα αυτό. Φυσικά είναι σημαντικό. Πρόεδρος. Και νομίζω ότι είπατε το 64% των επιδοτήσεων πηγαίνει στην αλία βυθόβιων ε, ηχθείων. Δηλαδή ο πελαγικός στόλος λαμβάνει μικρότερη επιδότηση και είναι λιγότερο αποδοτικός κερδοφόρος από βάση της ερευνάς και λαμβάνει μικρότερες απαλλαγές για τα καύσιμα, φορολογικές απαλλαγές. Γιατί το παραδείγματο χάρη, κάποια κράτη-μέλη έχουν μερική απαλλαγή για τους ε, στόλους ε, μακρινών αποστάσεων. Φαίνεται να υπάρχει λοιπόν ανισότητα μεταξύ των διάφορων τμήματων του στόλου. Okay. It's really... Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, όπως σας είπα, για την ανάλυση των δεδομένων να λάβουμε υπόψη μας ε, τους δια, τις διάφορους τομείς. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι τομείς παρόντες σε όλα τα κράτη. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι διάφορες χώρες εκτιμούν και συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά πράγματα στις ε, ε, άμεσες εισοδηματικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, εάν κάποια χώρα ε, έχει φορολογική ελάφρυνση που είναι τεράστιο ποσό και αυτό το συμπεριλάβει στην άμεση εισοδηματική επιδότηση, ενώ μια άλλη χώρα που δεν έχει ας πούμε ε, τράτες, ε, δεν, συμπεριλαμβα... δεν συμπεριλαμβάνει αυτές τα γρήγορα, δεν έχει γρηγρή ας πούμε, τα... Ε, δεν συμπεριλαμβάνει στις επιδοτήσεις, τότε προφανώς είναι κάπως τρευλωμένα τα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτά είναι, είναι θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν με μεγαλύτερη ανάλυση, περισσότερα στοιχεία, πιο κατακαιρματισμένα στοιχεία, με καλύτερη ερμηνεία όλων των ε, στοιχείων, των παραμέτρων που μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι όλα αυτά τα αποτέλεσματα πρέπει να, εξετασ... να αντιμετωπιστούν με μεγάλη σύνεση και προσοχή. Ωραία, ευχαριστώ. Α, η κυρία Λόβεν θέλει το λόγο πάλι. Ναι, έχουμε χρόνο. Και χρόνο και ενδιαφέρον το θέμα, γιατί να με υποφιληθούμε. Κοίταγα τον πίνακα 4 για την αποδοτικότητα. Δώσατε κάποια παραδείγματα για κατηγορίες ε, στόλου, για τις άμεσες εισοδηματικές επιδοτήσεις, ε, όπου βλέπουμε ε, μεγάλες αυξήσεις του ακαθάριστη, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Στην Πολωνία είχατε, έχουμε ε, μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο, στα ποσά από την, ε, ε, αν λάβουμε υπόψη μας τις άμεσες επιδοτήσεις ή όχι. Επίσης, για μια άλλη πολύ αμφιλεγόμενη αλληλευτική πρακτική, το περιθώριο αυξάνεται σημαντικά. Η αποδοτικότητα μάλλον αυξάνεται σημαντικά με τις ε, επιδοτήσεις. Κοιτάξτε, αυτό θεωρούσα ότι ήταν κάτι σημαντικό και έχω μαζί μου τον πίνακα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν πληροφορίες. Για την Πολωνία δεν συμπεριλαμβάνεται, όμως ξέρουμε ότι πάρα πολλά χρήματα δαπανήθηκαν για την απόσυρση πλοίων. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Γιατί αυτό το οποίο κάνουμε, και όπως είπε και ο κ. Μάρτισον, είναι ότι εμείς συλλέγουμε τα στοιχεία που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη και μετά κάνουμε κάποιους ελέγχους μένα, αλλά για να ε, ελέγχους όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων, γιατί μας δίνουν ας πούμε ε, στοιχεία σε, διαφόρου, σε διάφορους πίνακες που όταν κάνουμε την άθροισμα, το άθροισμα δεν μας βγαίνει ας πούμε. Γι' αυτό εμείς θέλουμε κάτι λογικό. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε από την αρχή είναι, τουλάχιστον, είναι να πάρουμε τα στοιχεία που μας δίνουν. Αυτό έχουμε σαν ε, πρώτη ύλη αν θέλετε. Επομένως για το Ηνωμένο Βασίλειο δυστυχώς δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί δεν το έχουμε εδώ. Κυρία Λόβεν, άρα χρειαζόμαστε εναρμόνιση στην, ε, ε, στα στοιχεία που δίνουμε για τις επιδοτήσεις. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό γιατί το αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής ε, για το μέλλον της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία ανάμεσα όλα τα κράτη-μέλη για στο τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις άμεσες ισοδηματικές επιδοτήσεις και τι όχι. Π.χ. οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν, όπως επίσης και οι επιδοτήσεις για την μόνιμη πάυση αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν, να μην συμπεριληφθούν και όλα τα άλλα να συμπεριληφθούν είναι μεγάλη συζήτηση που κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα θέματα. Και υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που προσπαθεί να καταλάβει τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και τι δεν θα πρέπει ανάλογα με τους κανονισμούς. Εγώ σαν επιστήμονας θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε είναι όλα τα στοιχεία λεπτομερώς ε, για να μπορούμε να κάνουμε τις ανάλυσεις μας, να πούμε το μακαθάριστο κέρδος, ε, ε, από εδώ αποκλείουμε κάποια πράγματα όταν το υπολογίζουμε το ακαθάριστο κέρδος. Ε, για να ορίσουμε το καθαρό κέρδος πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες όμως και εναρμονισμένες πληροφορίες αν θέλετε από πλευρά κρατών μελών. Διότι αλλιώς δεν μπορούμε να δώσουμε και δεν, στοιχεία, στοιχεία συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Άγχελ Κάλβο Σάντος ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, διαπιστώνουμε, να διαπιστώσω ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Κέντρο Ερευνών και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής είναι γνωστά σε εμά. Θέλω να τονίσω ότι χάρη στην προσπάθεια της Κομισιόν και των επιστημόνων, Έχουμε τώρα ένα σύνολο κοινωνικονομικών δεδομένων. Αυτό δεν ίσχυε πριν 10 χρόνια. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο λοιπόν ε, στο επίπεδο αυτό έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και τέτοιες μελέτες. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα για βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και ιδίως ε, τα δεδομένα για τις επιδοτήσεις. Όπως είπε και η συνάδελφος, ε, υπάρχει τώρα μία συζήτηση στην Οικονομική και Επιστημονική Επιτροπή Αλίας για να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τα δεδομένα σχετικά με τις επιδοτήσεις. Αυτό είναι ένα καθήκον που εκκρεμεί και ελπίζουμε να επιληθεί το επόμενο έτος. Επίσης, είναι σημαντικό όταν ερμηνεύουμε τα δεδομένα να έχουμε κατά ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση τα δεδομένα αυτά βασίζονται εν μέρη σε αναλύσεις του ΟΣΑ και αυτή η ανάλυση του ΟΣΑ αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως ε, προσεκτικοί απέναντι στα δεδομένα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω και υπόθηκε από τους συναδέλφους είναι ότι η συνεισφορά της αλίας ε, σε απόλυτη αξία κυμαίνεται γύρω στο 0,2% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως αναγνωρίζετε στη μελέτη και όπως ολίασαν οι συνάδελφοι, ο έμεσος αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεν δίνεται ο αριθμός αυτός στη μελέτη, αλλά πιθανότατα ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτινσον και την ε, κυρία Μπορέλο για την εξαιρετική τους παρουσίαση. Ξέρω πως δεν είχατε σχεδόν καθόλου χρόνο και ήταν πολύ δύσκολο, όμως ε, η συζήτηση που είχαμε μετά από την παρουσίασή σας αποκάλυψε το πόσο πολύπλοκο είναι το σύστημα και ελπίζω στο μέλλον να το επανεξετάσουμε. Γι' αυτό αν έχετε χρόνο για να κάνετε περισσότερο ενδελεχή έρευνα και να λάβετε στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα η Ελλάδα δεν συμμετείχε για, τους, για προφανείς λόγους, στο ζήτημα αυτό της κερδοφορίας. Ήταν καλό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη δουλειά σας. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πληροφορούμαστε από εσάς για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε. Προχωράμε τώρα στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης, τα διάφορα. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ. Ένα σχέδιο ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ζητήσαμε να μπει το, η πρόταση ψηφίσματο στην ε, μερίσια διάταξη Ολομέλειας του Δεκεμβρίου και ο λόγος είναι η αργοπορία της Λιθουανικής Προεδρίας σε, στις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο αυτό για παράδειγμα αναθεωρημένη εντολή θα συζητήσετε και θα συμφωνιστεί την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά τα άρθρα 26 έως 79. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο και αυτή η δυνατότητα έχει ήδη συζητηθεί με όλους τους κοιόδης συζητητές στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα πριν τον ε, τελευταίο τριμερή διάλογο υπήρξε συνένεση ανάμεσα στους κοιόδης εισηγητές. Η απόφαση λοιπόν να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου πρέπει να ληφθεί και να εγκριθεί από αυτήν εδώ την Επιτροπή έτσι ώστε η Γραμματεία να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ρωτήσω καταρχάς εάν μπορούμε να λάβουμε μια τέτοια απόφαση. Όχι. μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε μια συνένεση εδώ ότι εσείς συμφωνείτε να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερησία διάταξη της Ολομέλειας έτσι ώστε να πιέσουμε το Συμβούλιο. Κύριε Άγνιου. Ε, πρόεδρε, είναι καθήκον μου να μην επιταχύνω την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος, συμφωνούμε λίγο πολύ ομόφωνα εκτός από τον κύριο Άγνιου. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Το τελευταίο θέμα που έχουμε στα διάφορα είναι μία αναφορά, μια έκθεση όσον αφορά τα πολιτή σχέδια της ομάδας δράσης. Συναντηθήκαμε σήμερα το πρωί με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν και συμφωνήσαμε να εγκριθεί η πρώτη ενδιάμεση έκθεση βάσει της οποίας η Κομισιόν θα συντάξει και θα προετοιμάσει τα πολυετή σχέδια για, τα, για ορισμένα ε, είδη βασισμένοι στα κριτήρια που έχουν ήδη συζητηθεί και συμφωνηθεί και ελπίζουμε τα πρώτα τέτοια πολυετή σχέδια να συμφωνηθούν όταν θα έχουμε και την ε, συμφωνία από το Συμβούλιο. Η κυρία Φράγκα έχει κάτι να πει. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν συνέχισε αυτή η task force ε, ε, όπως λέγεται. Και ακριβώς αναφέρομαι στο θέμα της απόφασης για το Harvest Control Rule, για τον κανόνα ελέγχου της αλίευσης. Να σας πω ότι το έγγραφο που συζητήσαμε και συμφωνήσαμε σε επίπεδο διοργανικής συμφωνίας <laughs> είναι τόσο αμφίσιμο και τόσο αποδυναμωμένο που δεν μπορεί να πλήξει κανέναν. Θα ήταν θαύμα αν τώρα η Κομισιόν παρουσιάσει ένα πολιετές σχέδιο ακόμη και για ένα απόθεμα που να είναι τόσο αποδυναμωμένο που να περάσει την έγκριση του Συμβουλίου. Είναι συμβολικό σας λέω, γιατί έχει συμφωνηθεί από τα τρία όργανα και είναι η πρώτη τέτοια συμφωνία για τα πολιετή σχέδια που έχουμε δει στα πέντε έτη. Και επομένως ε, είναι ένα building block. Θα περάσουμε τώρα στην ελληνική προεδρία και έχουμε τρεις μήνες μέχρι το Μάρτιο για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στις πλέον πολύπλοκες συμφωνίες για τα ελεγκτικά μέτρα, για την νυχτά ήδη αλίας. Θα είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε σε αυτό. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μόνο στο πρώτο στάδιο, απλώς σας ενημερώνω. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 20 της ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Να σας πω ότι έχουν αποσταλεί συστάσεις από τη Γραμματεία και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε πως εγκρίνονται. Η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης, 16 Δεκεμβρίου, από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα και 17 Δεκεμβρίου από τις 9 έως τις 12.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε το δεκεμβρη Thanks. See you.